μιλάει για τον επεκτατισμό αυτό του προπολογισμού, για τα μεγάλα γραφεία. Πάμε στην Ινδονησία, στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω εγώ πού. Κοίταξα το χάρτη την τελευταία φορά. Τι φέρνει στην έκθεση αυτή το Συμβούλιο. Παραπάνω εκατομμύρια, τα οποία εξοδεύονται σε προπαγάνδα, σε κέντρα ευρωπαϊκής εμπειρίας. Ε, επίσης ε, νοικιάζουμε 15 νέα γραφεία και διάφορους managers. Περισσότερα χρήματα επίσης για την επίπλωση των γραφείων των Ευρωβουλευτών που την τελευταία φορά που κοίταξε ήταν μια χαρά. Και ερχόμαστε και στο Brexit. Και εδώ διάφορε επιλογέ αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Βέβαια, γιατί όχι. Ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί στο Westminster δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν κατά πόσο θα υλοποιήσουν τελικά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο. Κι όμως το 2014 εκλέχτηκαν οι ευρωβουλευτές, ε, δόθηκε εντολή με τις εκλογές του 2015 να γίνει δημοψήφισμα του 2016 και το αποτέλεσμα ήταν Brexit. Και το 2017 όντως εφαρμόστηκε, είπαμε ναι, ξεκινάμε για το Brexit. Και τώρα ποιος φταίει για όλα αυτά. Οι πολιτικοί στο Westminster τελικά αγνοούν την εντολή που έχουν πάρει και δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν. Εντάξει, αυτοί φταίνουν, όχι εσείς. Μεγάλη ανακούφιση, κύριε Άρνοτ. Δέχεστε μια ερώτηση από τον κύριο Ρούμπικ. Κύριε Ρούμπικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ξέρουμε όλοι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας και η συνθήκη της Ρώμης πάντα απαιτούν ομοφωνία για το θέμα του της έδρας και η έδρα είναι το Στρασβούργο. Γιατί η έδρα Στρασβούργο αμφισβητείται. Συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε εδώ και νομίζω ότι έχει απόλυτα έννοια. Για το Brexit βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα αποφασιστεί ε, σκληρό Brexit και χάος σε μερικές ώρες. Η Βουλή των Κοινοτήτων δεν έχει πάρει καμία απόφαση. Και θα μας ενδιέφερε να μας πείτε πώς θεωρείτε ότι θα ε, ε, καταλήξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύσκολο να απαντήσει κανείς σε μια ερώτηση που δεν έρχεται με ερωτηματικό. Σίγουρα συμφωνώ. Επικρατεί χάο στο Westminster τώρα και περιμένουμε οι πολιτικοί εκεί στη Βουλή των Κοινοτήτων να λάβουν αποφάσει και να ηγηθούν όσον αφορά το Brexit το οποίο ψήφισαν οι άνθρωποι, όσον αφορά το τσίρκο αυτό που ταξιδεύει μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου. Είναι απλώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σύστημα έχει χαλάσει, έχει καταρρεύσει. Το κοινοβούλιο δεν έχει κανέναν τη βασική δημοκρατική εξουσία που μπορεί να συνεδριάζει. Οπότε έχει καταρρεύσει το σύστημα αυτό που μπορεί να αποφασίσει το κοινοβούλιο. Κύριος Αρτουή έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοκρατία κοινοβουλευτική δεν έχει τίμημα, αλλά κοστίζει και εμείς τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε τη χρήση, την αυστηρή χρήση, τη μετρημένη χρήση των ευρώ που τίθεται στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να αποτίσω φορό τιμής στον Βλαντιμίρ Μάνκα που προετοίμασε την όλη ανάλυση του σχεδίου προπολογισμού για το Κοινοβούλιο. Το έκανα αυτό με προσοχή, με αυστηρότητα, με συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές. Χαιρετίζω την προσπάθεια που κατέβαλαν και την έξοχη ποιότητα της δουλειάς τους. Να σας πω ότι αυτή η αυστηρότης όσον αφορά τη διαχείριση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου ε, επηρεάζει και, το, και τις αρχές του Κοινοβουλίου και το κύρος του Κοινοβουλίου όταν έχουμε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο την περίοδο που ακολουθεί την ψηφοφορία του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η ψήφο που εκφράζουμε εδώ είναι προσωρινή ψήφο που θα επιβεβαιωθεί, θα κυρωθεί στην ψηφοφορία μα του μηνό Οκτωβρίου. Τούτων λεχθέντων. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα την εντύπωση που έχω σχηματίσει. Ότι θα πρέπει οι να διαλυθούν. Εδώ και πέντε χρόνια προεδρεύω τη Επιτροπή Προπολογισμών και κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια δυσκολία, διότι εξετάζουμε ένα σχέδιο προπολογισμού που αντικατοπτρίζει μια πολιτική που αποφασίζει το Προεδρείο και έπρεπε να εκφράσουμε αμφιβολίες ερωτηματικά όσον αφορά ε, τη στελέχωση, όπως τη δημιουργία θέσεων ε, εργασίας, ε, την διπλωματική εκπροσώπηση σε κάποιες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις που μας δόθηκαν δεν ήραν πάντοτε τα ερωτηματικά μας. Ε, πρόκειται όμω περί αποφάσεως του Προεδρείου και αποφασιών των ομάδων, οπότε στην πράξη δεν είχαμε τη δυνατότητα να αμφισβητήσουμε αυτέ τι επιλογέ. Πιστεύω συνεπώ ότι στην επόμενη θητεία θα πρέπει αυτή η αμφισημία να αρθεί όσον αφορά ε, τις διάφορες πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τα, χρήματα που περισσεύουν, εκεί που υπάρχουν υπερεκτιμήσεις των κονδυλίων που χρειάζονται και υπάρχει ε, χρήμα που έχει χρησιμοποιηθεί για τα ακίνητα. Πρέπει να υπάρχει αναθεώρηση όσον αφορά την πολιτική για τα ακίνητα, για τα κτίρια. Και θα πρέπει να είναι ειλικρινή ο προπολογισμό όταν καταρτίζεται. Από τι αφορά τιμή όλου εκείνου που διαδοχικά υπήρξαν εισηγητέ για το σχέδιο προπολογισμού του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ του και όδη εισηγητέ, αναγνωρίζω την προσπάθειά του και εκφράζω το θαυμασμό μου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ένα συνάδελφο είναι στη δικασία Catch the Eye, ο κύριος Καστάλντο. Κύριε Καστάλντο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δυστυχώς θεωρώ ε, ότι να βλέπω και ε, αλλαγή του προπολογισμού τον επόμενο χρόνο ένα χρόνο όπως αυτό να υπάρχει αλλαγή, όπου υπάρχει δυνατότητα του Brexit, όπου αυτή η λύση μπορεί να χάσουμε 46 έδρες εκπροσώπου. Παρ' όλα αυτά τη βλέπουμε μια αύξηση των δαπανών στην πρόβλεψη. Στα, στα του, προ, του Προεδρείου εξέφρασα άποψη κατά των πρωτοβουλειών, όπως τα νέα, τα νέα γραφεία εκπροσώπησης ε, του Κοινοβουλίου, που είναι πολύ δαπανηρά γραφεία, και άλλες αποφάσεις για την αναδιάθρωση του, ε, του PHS, του κτηρίου. Και μετά τεράστιε δαπάνε που σχετίζονται με την τριπλή μα έδρα που εξακολουθεί να είναι το σύμβολο μια έλλειψη ε, σεβασμού έναντι των χωρών εκείνων από τα οποία ζητούμε πάντα μεγαλύτερε θυσίε αυστηρότητα και λιτότητα. Ένα δισεκατομμύριο για τα επόμενα πέντε χρόνια θα κοστίσει αυτή η τριπλή έδρα. Και κλείνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ ε, να πω ότι 370 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη θητεία για κόμματα και ιδρύματα. Αστρονομικά ποσά δικαιολόγητα προβλέπονται και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε, σύντομα θα μα ζητήσουν το λόγο να δώσουμε λογαριασμό για αυτά τα αστρονομικά ποσά. Συνάδελφοι, η συζήτηση περατώθηκε και ψηφίζουμε την έκθεση αύριο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι έκθεση Μισελ Ντατέν, η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Καλωσορίζουμε τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο και, του δίνουμε, και δίνουμε λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά, στον κύριο Ταντέρ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι Σκιώδης, συνάδελφοι, εδώ και 40 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Στις χώρες μας έχει υπάρξει ουσιώδης πρόοδος. Η νομοθεσία αυτή αναθεωρήθηκε πριν από 20 χρόνια ακριβώς και τώρα χρειάζεται μια περαιτέρω αναθεώρηση για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της επιστημονικής πρόοδου που έχουν μεταφραστεί σε νέες προδιαγραφές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Αλλά πρέπει, όπως μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εντάξουμε και τις προόδους της γνώσης όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, όπως ε, την παρουσιάζει η οδηγία πλαίσιο για το νερό και να λάβουμε υπόψη τι προσδοκίε των πολιτών για πρόσβαση στο νερό και στη διαφάνεια. Τον περασμένο Οκτώβριο, στην Ολομέλεια, ψηφίσαμε την έκθεση για την αναθεώρηση τη οδηγία. Η οδηγία αυτή, που κυρίω αναθεωρεί τι παραμέτρου, προτείνει μια νέα μέθοδο αξιολόγηση των κινδύνων που επιτρέπει να προλάβουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τους κινδύνους ε, ε, ρήπανση. Και θα θέσει το κοινό ενώπιον των ευθυνών του, θα έχουμε μια διαχείριση με βάση τους κινδύνους, τις παραμέτρους ποιότητας και την πρόσβαση στο νερό. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε νερό υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, ε, σε λογικό κόστος και με πλήρη διαφάνεια έναντι των Ευρωπαίων καταναλωτών, με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Και παρά την εργασία που χρειάστηκε να γίνει, το Κοινοβούλιο απέδειξε ότι είναι στο ύψος των ε, προσδοκιών των πολιτών και από τον Νοέμβριο ξεκινήσαμε τι διαπραγματεύσει και καταλήξαμε σε διοργανική συμφωνία πριν από το τέλος της θητεία. Δυστυχώ. η καθυστέρηση για την έγκριση του κειμένου στο Συμβούλιο δεν μας επιτρέπει σήμερα να θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι ικανοποιητική. Αντίθετα, είναι πολύ λεπτή η κατάσταση, γιατί δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να έχει ε, γίνει αντικείμενο διαπραγματεύση ε, από τριμερεί διαλόγους και να έχει ψηφιστεί. Χαιρετίζω τι προσπάθειες ε, της Ρουμανική Προεδρίας για να καλυφθεί καθυστέρηση μέσω της παρουσίασης γενικής προσέγγισης στις 5 Μαρτίου. Αλλά αυτό είναι αργά. Δεν έχει το Κοινοβούλιο επαρκές περιθώριο για να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσει πριν τι ευρωεκλογέ. Η έκθεση αυτή έχει και τεχνικό περιεχόμενο και πολιτικό περιεχόμενο και επιπτώσεις. Μετά την ψήφιση πρώτη ανάγνωση αύριο θα είναι η επίσημη θέση του Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και από εδώ και μπρο θα πρέπει η Φιλανδική Προεδρία να διαπραγματευτεί αυτό το κείμενο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης οι οποίοι με βοήθησαν στις προσπάθειές μου και ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Και τώρα καλώ τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή κύριο Νταντά και τους Κιώδης για τη σκληρή εργασία που επετέλεσαν για την πρόταση για μια αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου συμβαδίζουν με τις κύριες κατευθύνσεις της πρότασής μας. Παράλληλα, λυπάμαι, που λόγω της αργής πρόοδου στο Συμβούλιο δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει διοργανική συμφωνία πριν τις ευρωεκλογές. Υπενθυμίζω ότι κύριο στόχο τη πρότασή μα είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ποσίμου ύδατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 21ο αιώνα. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που σήμερα οι περισσότεροι πολίτε που ζουν στην Ένωση έχουν ε, πόσιμο νερό στη διάθεσή τους παγκοσμίω υψηλωτά του επίπεδου. Με την πρότασή μα θα διατηρήσουμε αλλά και περαιτέρω θα βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση με αυστηρότερες προδιαγραφές και πιο κατάλληλες οριακές τιμές. Την περασμένη εβδομάδα, στις 22 Μαρτίου, είχαμε την επέτειο της, ε, μάλλον είχαμε την Παγκόσμια ε, ημέρα για το Ίδωρ με σύνθημα «Κανείς δεν πρέπει να μην έχει πρόσβαση στο Ίδωρ». Η Ευρώπη, λοιπόν, είναι μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμού που δεν αφήνει κανένα κατά μέρο. Οι υποχρεώσει ε, μέσω τη αναθερμένη οδηγία να υπάρχει για τα πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού επαρκής πρόσβαση σε καθαρό νερό ακριβώς βασίζεται σε αυτό το όραμα. Είναι αποτέλεσμα της, πρώτη της πρώτης ε, επιτυχούς πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών για το δικαίωμα στο νερό που στηρίχθηκε από 1,8 εκατομμύρια συμπολίτες μας από παράδειγμα λοιπόν του πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Θα βελτιώσει η πρόταση την κατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων ε, ατόμων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρότασή μα για την πρόσβαση στο νερό είναι επίση ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια επίτευξη του στόχου 6 των ε, βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Και χαιρετίζω την πρόταση του Κοινοβουλίου να υπάρχει πρόσβαση για όλου στο νερό. Είναι σημαντικό αυτό εν ώψη των μελλοντικών συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών τη αρχή της νομοθετικής αρχής. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος αποφάσισε τη γενική προσέγγιση στις 5 Μαρτίου, όπου στο συμβαστικό κείμενο υπάρχει μια λεπτή ισορροπία με πολύ περιορισμένε προποθέσει για την πρόσβαση στο νερό. Κάποια κάτι μέλη, όντω, ήταν κατά η πρόσβαση στο νερό να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, γνωρίζω ότι εδώ η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ε, η εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών θέλει να υπάρχει αυτή η ρύθμιση και περαιτέρω η πρόταση του Συμβουλίου για το άρθρο 10α για τα υλικά σε επαφή με το νερό προκαλεί διάφορες ανησυχίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό ε, επιφυλασσόμεθα τις θέσεώ μας για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις αλλά δηλώνουμε ως Επιτροπή ότι θέλουμε να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε περαιτέρω τι ανησυχίε για αυτό το άρθρο. Και θα ενημερώσουμε του συνομοθέτε εν ευθέτω χρόνο για τα αποτελέσματα τη έρευνά μα. Σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται και θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και την επερχόμενη Φιλανδική και την μεθεπόμενη Κροατική Προεδρία για να ξεκινήσουν ε, όσο το δυνατόν ταχύτερα οι πραγματεύσει. Επίση, υπογραμμίζω ότι ως έντιμος διαμεσολαβητής αυτών των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, προωθήσει τους σημαντικούς στόχους αυτής της πρότασης που νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμεθα. Τέλος, υπενθυμίζω ότι το ασφαλές πόσιμο είδων είναι ουσιώδες για τους συμπολίτε μας. Οι λύσεις που προτείνουμε θα φέρουν θετικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν καλό το Κοινοβούλιο να στηρίξει την ε, φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύσουμε ακόμη περισσότερο την υγεία των συμπολιτών μας προτείνοντας αυστηρές προδιαγραφές υγείας και διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβασή τους στο νερό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Λίζε, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το πόσιμο νερό είναι το τρόφιμο που ελέγχεται καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι υποχρέωση για μας. Πρέπει ε, πάντα να ακολουθούμε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά το πόσιμο νερό ακόμα ασφαλέστερο. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Στη διαδικασία πάντα τονίσαμε ότι αυτά τα οποία αποφασίζουμε θα πρέπει να βοηθήσουν και τις μικρότερες εταιρείες υδάτων και όχι να υποφελθούν μόνο οι μεγάλες εταιρείες που προτείνουν νέες μεθόδους ανάλυσης. Ε, τελικά πρέπει όλα αυτά να είναι χρηματοδοτήσιμα. Γιατί σε τελευταία ανάλυση ο φορολογούμενος τα πληρώνει. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η ασφάλεια, αλλά το κόστος ιδιαίτερα για τις μικρότερες εταιρείες υδάτων, πρέπει να παραμείνει σε λογικό επίπεδο. Το μεγάλο θέμα είναι το θέμα της πρόσβασης στο νερό. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα το να υπάρχουν διάφορα σημεία στην Ευρώπη, όσο να τον περισσότερα, όπου να υπάρχει ε, δωρεάν πρόσβαση στο νερό σε διάφορου δημόσιου χώρου. Όσο να τον περισσότερου. Πολύ καλό στα καφέ, νύα και τα εστιατόρια, το πόσιμο είδωρ να παρέχεται δωρεάν. Αυτό είναι καλό για του συμπολίτε μα και θα στηρίξουμε έτσι και την πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε εξοικονομήσεις γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές το εμφιαλωμένο είδωρ ε, μεταφέρεται εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αυτό κοστίζει καύσιμα, δημιουργεί λοιπόν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν νομίζουμε ότι είναι και τόσο σκόπιμο να πίνουμε αυτό το εμφιαλωμένο νερό συνεχώς. Ε, το νερό της βρύσης είναι επίσης πολύ καλό. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, όλα που θεωρούμε εμείς ε, σωστά και καλές ιδέες δεν θα έπρεπε να αποφασίζεται κεντρικά και συγκεντρωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβάλλεται σε κάθε γωνιά της Ένωσης. Υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας. Γι' αυτό εμείς ως ΕΛΚ έχουμε την άποψη ότι ο συμβιβασμός που ε, βρέθηκε στο Συμβούλιο είναι πολύ καλός και νομίζω ότι πρέπει να τον προσεγγίσουμε στις ε, διαπραγματεύσεις. Να υπάρχουν κίνητρα, αύξηση της ε, ε, ευαισθητοποίησης. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους μας παρά να επιβάλλουμε σε όλους τους έχουν ένα καφενείο στην Ευρώπη τι θα πρέπει να κάνουν. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις αντιευρωπαϊκές διαθέσεις. Γι' αυτό στηρίζουμε την ιδέα, αλλά δεν πρέπει να είναι η νομοθεσία άκαμπτη. Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Μισελ Νταντά, Δυστυχώ δεν θα επανεκλεγεί, γιατί δεν θα είναι υποψήφιο, αλλά επέτυχε για πολλά θέματα, θαυμάσια αποτελέσματα, όπως αυτό αγαπητέ Μισελ, ευχαριστώ για την εργασία σου και καλή τύχη στο μέλλον. Ναι, και εγώ συμμερίζομαι όσο είπατε τα καλά σας λόγια του κύριου Δύο μισή λεπτά ο κύριος Πάλμερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Νταντάν, για το συντονισμό του και τις προσπάθειές του για το θέμα αυτό. Και ευχαριστώ πολύ και τους κοιόδης εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Επίσης, ευχαριστώ πολύ το προσωπικό, τους βοηθούς μας, που δούλεψαν μήνες τώρα ε, πάνω σε τόσο περίπλοκα ζητήματα για να καταλήξουμε σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Τώρα, πολλές οργανώσεις και διάφοροι φορείς ήρθαν σε επαφή μαζί μας όλους αυτούς τους μήνες και θέλω και αυτούς να τους ευχαριστήσω για τις προσπάθειές τους και για το ενδιαφέρον που έχουν δείξει. Όντως είναι τεράστιο το εύρος των φορέων που ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα που όντως είναι πολύ περίπλοκο. Οπότε τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξή τους που κάνουν εκστρατείες και συνεχίζουν να μας πιέζουν για να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων. Το κείμενο που έχουμε μπροστά μας είναι λοιπόν καλύτερο από ό,τι θα ήταν χωρίς τη δικιά τους βοήθεια και από αυτά που προτείναμε πέρυσι. Αυτό που είναι κρίμα, είναι κρίμα που το Συμβούλιο ε, πήρε τόσο πολύ χρόνο για να καταλήξει σε μία απόφαση και να μην μπορέσουμε νωρίτερα να μπούμε σε τριμερή διάλογο. Θα γίνει αυτό στην επόμενη θητεία. Τι να κάνουμε. Όποια και αν είναι η πολιτική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω να συνεχίσει να δείξει τη δέσμευσή του για το δικαίωμα αυτό στο νερό. Πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό το Κοινοβούλιο. Και εμείς ε, πρέπει να δούμε ότι αυτό που πετύχαμε με αυτή την έκθεση ήταν τεράστια πρόοδος και ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Οπότε το Συμβούλιο ε, δεν θα έπρεπε ή το νέο Κοινοβούλιο να μειώσει, να περιορίσει τις φιλοδοξίες αυτού του κειμένου γιατί μας, μας ενδιαφέρει φυσικά η τεχνολογία, η επιστήμη, όλα τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε το νερό να είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλές. Επίσης, ασχολούμαστε και με το βασικό ζήτημα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί δεν μπορεί να είναι δίκαιο σήμερα στον 21ο αιώνα να υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό είναι πολύ βασικό αυτό για μας τους ευρωβουλευτές σε αυτή τη θητεία. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτή ήταν η προσέγγιση της σοσιαλιστικής ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών μας πάνω σε αυτό το φάκελο. Και για μένα είναι τελευταία νομοθετική πρόταση ε, με την οποία μπλέκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελευταία νομοθετική πρόταση για μένα και χαίρομαι που είναι ακριβώς αυτή. Γιατί πρόκειται για μια οδηγία η οποία θα επηρεάσει τη ζωή και την καθημερινότητα όλων των Ευρωπαίων πολιτών κάθε μέρα της ζωής τους. Και δεν είναι πράγματα που πρέπει να παίρνουμε σαν δεδομένα, το καθαρό πόσιμο νερό δηλαδή. Το θέμα δεν είναι βρύση ή όχι βρύση, είναι ποιότητα, είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να πιέζει για το δικαίωμα αυτό σε καθαρό νερό. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος αυτή η έκθεση. Και όταν οι άνθρωποι τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, χρόνια ε, θα αναρωτιούνται τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού. Διασφαλίζει ότι όπου και αν βρισκόσαστε, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Στρασβούργο, στι Βρυξέλλε, οπουδήποτε αλλού, ανοίγετε τη βρύση και έχετε ποιότητα πόσιμου ύδατος. Ευχαριστούμε. Ένα μισή λεπτό τώρα, ο κύριος Χότ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το νερό είναι σημαντικότατο για το ανθρώπινο σώμα. Και είναι μια κληρονομιά σημαντική και για μας και για μελλοντικές γενιές. Δυστυχώς οι πόροι είναι περιορισμένοι. Και γι' αυτό χρειάζεται ορθή διαχείριση των υδάτων. Και πρέπει να κάνουμε και οικονομίες στο νερό. Τουλάχιστον 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό χάνονται και σπαταλιώνται σε μεγάλες πόλεις. Αυτό σημαίνει νερό που αφορά 10 με 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες οικονομίες. 900 λίτρα για κάθε τετραμελή οικογένεια. Κάθε χρόνο χάνουμε 20.000 λίτρα νερού εάν δεν κλείνουμε τη βρύση μας σωστά και στάζει. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται μια αυστηρότητα, μια προσοχή ε, όσον αφορά το νερό και επίσης και για παθογόνες ουσίες και για το μόλιβδο χρειάζονται ε, μέτρα και τα μικροπλαστικά και χρειάζεται και καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τμήμα ε, της νομοθεσίας αυτής. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι 600 εκατομμύρια ευρώ αν γίνουν όλα αυτά σωστά. Αυτό είναι κάτι που σχετίζεται και με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ε, το νερό πρέπει να ελέγχεται συνεχώς, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Επίσης χρειαζόμαστε και τη διάθεση δωρεάν νερού σε δημόσιους χώρους όπως και στα εστιατόρια ακόμα. Ε, χρειάζεται υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού. Πρέπει να θυμόμαστε το νερό σημαίνει νερό, σημαίνει ζωή. Επίσης, πάντα βλέποντας το διάστημα, το ανοιχτό διάστημα, πάντα ψάχνουμε το νερό και διαρωτώμαθα για το νερό. Αυτό είναι κάτι πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας το νερό. Είμαι πιο ευέλικτη απόψε, λέει ο Πρόεδρο. Παρακαλώ όμω ότι μην το παρακάνετε. Η κυρία Μούλερ, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή μα έκανε αυτή την πρόταση για την αναθεώρηση τη οδηγία για το νερό, αντιδρώντα στην πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, το δικαίωμα στο νερό. Το κόμμα μου, οι ελεύθεροι ε, ψηφοφόροι, είναι υπέρ τη ε, συμμετοχής ε, των ε, πολιτών στην πολιτική ζωή. Γι' αυτό μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις πρωτοβουλίε των πολιτών και να αντιδρούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά σε αυτές. Θεωρώ ότι εμεί, ω Κοινοβούλιο επίση δράσαμε αποτελεσματικά. Παρά τις τεχνικής, την τεχνική και πολιτική πολυπλοκότητα του θέματο, ήδη τον Οκτώβριο υποβάλαμε την έκθεσή μα. Ήμασταν διατεθειμένοι και έτοιμοι για να με το Συμβούλιο. Όμω το Συμβούλιο αντίθετα καθυστέρησε πάρα πολύ. Άρα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε την οδηγία πριν το τέλος της θητείας. Αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία. Γι' αυτό αύριο πρέπει να αποφασίσουμε για την έκθεση αυτή στην πρώτη ανάγνωση και θα στείλουμε έτσι ένα μήνυμα προς τους συμπολίτε μας ότι η συμμετοχή τους δεν είναι απλώς κενές λέξεις για μας, αλλά ουσιώδες. Η έκθεσή μας όμως και ε, περιέχει και πολύ καλές προτάσεις επί του περιεχομένου. Προτείνουμε μία λύση, ούτω ώστε στο μέλλον να αντιμετωπίζουμε τα μικροπλαστικά και άλλες ε, επιζήμιε ουσίες στο πόσιμο είδο. Έτσι θα υπάρχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα του πόσιμου ύδατος και κάνουμε και προτάσεις, ούτω ώστε να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους χωρί να δημιουργούμε προβλήματα σε ήδη υπάρχουσε δομέ όπως ε, την ε, παροχή του ύδατος που γίνεται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και γενικότερα στην Ήπεθρο. Ελπίζω αύριο να δοθεί σωστή διαπραγματευτική εντολή για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή Μισελ Νταντάν για την πολύ καλή συνεργασία και τους σκιώδης. Το πόσιμο νερό είναι το τρόφιμο που έχουν γίνει οι περισσότερες έρευνες και ο καθένας μας μπορεί να πιει νερό της βρύσης άφοβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Γιαβόρ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το υγιές πόσιμο νερό είναι βασικό δικαίωμα. Και κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει δικαίωμα σε αυτό. Και γι' αυτό το δικαίωμα στο νερό, η πρωτοβουλία των πολιτών, αυτό αφορούσε το δικαίωμα στο νερό. Και ήταν ε, η πρώτη πρωτοβουλία ευρωπαϊκή πολιτών που ήταν επιτυχής είπε αυτά που έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή τη βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση και ελπίζουμε να την υποστηρίξει αύριο στην πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά τα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκέ πόσιμο νερό, διότι είναι μέλη μειονοτήτων, έχουν αποκλειστεί, έχουν περιθωριοποιηθεί από την κοινωνία και γι' αυτό δεν έχουν πρόσβαση στο κατάλληλο πόσιμο νερό. Μιλάμε για εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί διάφορε κυβερνήσει, όπω η Ουγγρική κυβέρνηση, δεν μπορούν να εγγυηθούν την αναγκαία σωλήνωση του ώστε να φτάσει το νερό σε αυτού του ανθρώπου και να πληρούνται οι απαραίτητε προποθέσει που προβλέπουμε για ε, το υγιεινό πόσιμο νερό. Δεν μπορούν να το εγγυηθούν αυτό παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό, υποστηρίζοντα τα κράτη-μέλη, εξασφαλίζοντα ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα που θα επιτρέπουν σε όλου να έχουν πρόσβαση στο καλό νερό. Οι πόροι δεν χρησιμοποιούνται σωστά δυστυχώ ε, και τελικά διασπαθίζονται τα ποσά, πηγαίνουν στη διαφθορά και τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο έχουν προσημειωθεί. Δηλαδή να υπάρχει εγγύηση για πόσιμο νερό υψηλή ποιότητα. Το πόσιμο νερό υψηλή ποιότητα δεν σχετίζεται μόνο με την υγεία και την ασφάλεια, όπω αναφέραμε στη συζήτηση. Εάν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ε, έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτε στο πόσιμο νερό από τη βρύση, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη ζήτηση για το εμφιαλωμένο νερό. Και αν μειωθεί επαρκώ η μείωση για το εμφιαλωμένο νερό, τότε θα μειωθεί δραματικά και ε, το επίπεδο των αποβλήτων. Θα πρέπει να αποκτήσει ο κόσμο εμπιστοσύνη στο πόσιμο νερό τη βρύση. Και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση. Δυστυχώ το Συμβούλιο δεν έχει κάνει τη δουλειά που έπρεπε να γίνει πάνω στο θέμα. Και στο μέλλον, όχι μόνο το Συμβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη που συνεδριάζουν στο Συμβούλιο που να κάνουν τα πάντα του να εξασφαλίσουν ότι αυτέ οι προτάσει εφαρμόζονται σωστά και ότι κάθε Ευρωπαίο πολίτη έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μπόιλαν. Ευχαριστώ, αγαπητοί συναδελφοί. Όσοι έχουμε εργαστεί με το κίνημα για το καθαρό είδωρο, απογοητευόμαστε σήμερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να αντιμετωπίσει το θέμα. Δεν τα καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζητούν οι πολίτε. Πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Και γιατί, γιατί το ανθρώπινο δικαιώματα για το είδωρ είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο και τόσο δύσκολο. Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε αυτοί που εκπροσωπούμε απευθεία τον κόσμο. Και όμως τους αδικούμε μετά από τη δικιά τους πρωτοβουλία που μάζεψε τόσα εκατομμύρια υπογραφές. Είμαστε πίσω στη θέση του 2015. Εμείς δυσκολευόμαστε να εγκρίνουμε αυτήν την νομοθετική πρόθεση, γιατί, πρόταση, γιατί αν την εγκρίνουμε είναι σαν να προδίδουμε τον κόσμο που ζήτησε καθαρό νερό. Η πρωτοβουλία ε, ζητούσε καθαρό είδωρ για 2 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχουν και ζητά καθολική πρόσβαση στο νερό με προσιτές τιμές. Όμως καταλήγουμε στους στόχους φιλελευθεροποίησης και για το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα του κόστους, της απόδοσης, έτσι όμως ξεχνάμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι αρκετό και δεν ανταποκρίνεται στα όσα ζήτησαν με την πρωτοβουλία τους οι πολίτες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Συνάδελφε Μπόιλαν, υπάρχει γαλάζια κάρτα. Μία ερώτηση θέλω να σας υποβάλω. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα για σας. Συνάδελφε Ρούμπικ, την ερώτησή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Μπόιλαν. Βεβαίω είναι σημαντικό το νερό να δίδεται και δωρεάν. Το νερό είναι ένα κοινό αγαθό, αυτό είναι αυτονόητο. Και αυτή την προσέγγιση πρέπει να την ακολουθήσουμε αποφασιστικά. Αλλά είναι το θέμα των υποδομών μέσω των οποίων παρέχεται το είδωρο. Η υποδομή πρέπει να πληρώνεται, έχει ένα κόστος. Θεωρείτε ότι είναι καλή μέθοδος στο μέλλον η υποδομή αυτή να είναι ε, ιδιοκτησία του δημοσίου του ώστε να έχει την καλύτερη τιμή ο καταναλωτή. Συνάδελφε Μπόιλαν, την απάντησή παρακαλώ. Οι χώρες μέλη έχουν την αρμοδιότητα να διαχειριστούν αυτό το θέμα. Και εμείς έχουμε τεράστια προβλήματα στην Ιρλανδία, επειδή ακριβώ παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικά μας συστήματα. Εμεί έχουμε μηδενική φτώχεια για το είδωρο στην Ιρλανδία. Και γιατί, γιατί εμεί πληρώνουμε με την φορολογία και όχι ε, να τιμωρούμε τον κόσμο όταν δεν έχει χρήματα να πληρώσει νερό. Όχι, δεν θέλουμε αυτήν την ελευθέρωση των υποδομών ε, του νερού. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά, κύριε Εύη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ιταλία το νερό σαν κοινό αγαθό είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζητήσεως χάρη στο κίνημα των πέντε αστέρων που στο Κοινοβούλιο έχει καταθέσει νομοθέτημα ε, ξανά νομοθέτημα μετά το 2011, 8 χρόνια μετά για το νερό. Η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε των πολιτών όσον αφορά το πόσιμο νερό. Για λόγω των χωρών τη Κεντρικής Ευρώπης που για μήνε στο Συμβούλιο δεν έκανα καμία αναφορά στην, στο πόσιμο νερό, στο πόσιμο νερό. Αναγκαστήκαμε να ξαναψηφίσουμε το ε, κείμενο που τον περασμένο Οκτώβριο ψηφίστηκε το Κοινοβούλιο. Και το αναθέτουμε στην επόμενη θητεία για τι επικείμενε διαπραγματεύσει. Κατά την άποψή μα όμω αυτό είναι κακή πρόταση διότι οι συνάδελφοι της μεγάλης πλειοψηφίας συντηρητικής του Κοινοβουλίου ε, έκλεισαν την, τα, τα μέτρα όπως το, ε, την καλύτερη πρόσβαση στο είδον όπως το δικαίωμα που είναι όλων και πώς ε, μπορεί να εφαρμοστεί σωστά το right to ε, water. Υπάρχει και ευθύνη διότι αρνήθηκε να είναι μηδέν το όριο για τις ε, φθοριούχες ουσίες. Τι ουσίε ΦΑΣ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία που τέθεται σε ισχύ και που χρονολογείται από το 1998. Με πονίδιστο τρόπο έχετε θεσπίσει διαφοροποιήσει επικίνδυνε για τα διάφορα χημικά αυτή τη οικογένεια χημικών και κάποια φάστα θα μπορούσαν να γίνουν ανεκτά σαν ουσίε και δεν καλύπτονται νέα οδηγία για το πόσιμο νερό. Αλλά είναι σαφέ ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και αυτό σημαίνει στην περιοχή του Βένετο δείχνει προφανώ ότι καμία από αυτέ τι τοξικέ ουσίε δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκεται μέσα στο πόσιμο νερό και ούτε να σωρεύεται στο αίμα των παιδιών μα για το συμφέρον των Ιταλών και Ευρωπαίων πολιτών, για το συμφέρον αυτών. Ελπίζω επαντήστε το πόσιμο νερό να φτάσουν σύντομα και αναθεώρηση ε, που πρέπει να γίνει για να έχουμε τη σωστή ποιότητα πόσιμου νερού, να είναι κάτι που μπορεί να γίνει μαστηρότητα αυστηρότητα χωρί να υπάρχουν ε, ε, υποχωρήσει ενάντια τη βιομηχανία και να γίνει δελεχή ανάλυση όσον αφορά τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν για την πρόσβαση στο πόσιμο νερό ποιότητα. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λεπρετών. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πόσιμο είδωρ είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί πράγματι έχω ασχοληθεί με το νομικό καθεστώ του ύδατο και έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου στο Πανεπιστήμιο πριν από 70 χρόνια. Πρόκειται για οδηγία που ξεκίνησε από το 88 και σήμερα πάλι με το θέμα του ύδατο κλείνονται στα σταδιοδρομία μου εδώ είχαμε δύο εκατομμύρια υπογραφές στην πρωτοβουλία των πολιτών που ζητούσαν πρόσβαση στο είδωρ όλων των ευάλωτων ομάδων και των Ρωμά. Ο στόχος είναι ευγενής, αλλά υπάρχει και επικουρικότητα η ρύθμιση για το νερό είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι, οι διαταράκτες, οι ενδοκρινικοί ή τα πλαστικά ε, ρηπαίνουν το νερό, οι χώρες μέλη πρέπει να δράσουν αφού συνονοηθούν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Βρυξελών. Όσο για την καθολική πρόσβαση στο νερό, οι χώρες μέλη μπορούν κάλλιστα να διασφαλίσουν την πρόσβαση αυτή χωρίς να χρειάζονται μαθήματα ηθικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα μην είμαστε χαζοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χειραγωγήσει την κατάσταση των Ρωμά ώστε να αποκτήσουν καινούριε αρμοδιότητε για τέτοια θέματα. Η Ευρώπη των Εθνών, που θέλω εγώ, πρέπει να αντισταθεί σε τέτοιου χειρισμού, ώστε να επιστρέψει στα κράτη η πραγματική κυριαρχία του, το δικαίωμά του. Σα ευχαριστώ, κυρία Γιούζο. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει αναθεώρηση της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα για το πόσιμο είδωρ και πιστεύω ότι είναι καλές οι προτάσεις αυτές γιατί σήμερα έπρεπε όντως να υπάρξει αναθεώρηση και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να εντοπίσει τέσσερις τομείς που πρέπει να ε, βελτιωθούν. Είναι οι παράμετροι, είναι η προσέγγιση βάση κινδύνου, είναι η διαφάνεια και η πρόσβαση σε πληροφορίε και τελικά έρχονται σε επαφή με το νερό. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι χώρε μέλη εφαρμόζουν τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το πόσιμο είδωρ αρκετά καλά. Τώρα κάνουμε ένα παραπάνω βήμα προ τα μπρο που θα μα επιτρέψει να προλάβουμε προβλήματα. Τώρα έχουμε βελτιώσει τις τεχνικές μας γνώσεις, έχουμε νέες τεχνολογίες και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τις ε, περιβαλλοντικές μεταβλητές. Έτσι βελτιώνεται η οδηγία για το είδωρ. Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία βελτίωσης όσον αφορά την πρόσβαση σε πόσιμο είδωρ ποιότητας, όσον αφορά την ε, κατανάλωση του ύδατος, όσον αφορά τις πηγές ύδατος, πολύ σημαντικό, όσον αφορά την πρόληψη των ε, επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και φροντίζει και για την ε, καλύτερη προστασία από διάφορα υλικά. Προσφέρει επίσης λύσεις για το νερό σε πλαστικά μπουκάλια. Επίσης, οι μικροί διανομής ύδατος έτσι μπορούν να έχουν περισσότερη ευελιξία από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Τέλος, συγχαίρω ειλικρινά τον συνάδελφό μου, τον δόκτωρα Νταντάν, για το έργο του που βοήθησε για την βελτίωση της οδηγίας αυτής και φρόντισε επίσης και για το θέμα του κόστους. Λυπάμαι που δεν υπήρξε αρκετή ευέλιξή από πλευρά του Συμβουλίου για να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκούτελαντ. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό αν διψούν. Και αυτό το νερό πρέπει να είναι ασφαλές. Ασφαλές προς πόσιν. Και αυτό ισχύει για όλους. Είτε κάποιος έχει σπίτι ή δεν έχει σπίτι, είτε ανήκει σε κάποια πλειοψηφία, σε κάποια μειονότητα ή αεροκατοικημένη περιοχή της υπαίθρου ή σε κάποια κοσμοπολίτικη πόλη. Αλλά μέχρι τώρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό ασφαλές πόσιμο νερό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το νερό που πίνουμε πρέπει να είναι ασφαλές. Δεν μπορεί να υπάρχουν επικίνδυνα χημικά σε αυτό το νερό που να απειλούν την υγεία μα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε συνεπώ τι προδιαγραφέ μα, τι οριακέ τιμέ επίση και αυτέ πρέπει να βελτιωθούν και η ανθρώπινη υγεία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών. Οι ενδοκρινικοί διαταράχτε πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι είναι ουσίε που οδηγούν σε διαβήτη, σε άλλε επικίνδυνε ασθένειε επίση ή προβλήματα αγωνιμότητα συμβάλλουν σε όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να γίνει για να μην έχουμε τέτοιες επικίνδυνε ουσίε το πόσιμο νερό μα στο Κοινοβούλιο. Έχει μια ισχυρή εντολή, ισχυρή διαπραγματευτική θέση σε αυτό το τομέα και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη που θέλουν να χαλαρώσουν οι κανόνε. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να σταθεί και να υπερασπιστεί την υγεία των ανθρώπων και το δικαίωμά μα σε καθαρό υγιεινό νερό. Στις διαπραγματεύσεις όμως θα πρέπει να ακούσουμε να δούμε ποια η κατάσταση επικρατεί διάφορες χώρες. Υπάρχουν γεωγραφικές διαφορές, πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού. Γι' αυτό η θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχει κάποια ευελιξία που θα την παρέχει στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε η καλύτερη λύση, η πιο πρακτική λύση να επιλέγεται κάθε φορά σε κάθε περίσταση. Το καθαρό νερό είναι κάτι το οποίο είναι δικαίωμα όλων. Συνάδελφοι και έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η κατανάλωση ύδατος είναι έξι φορές παραπάνω από ό,τι ήταν πριν από 100 χρόνια και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό που περιμένουμε είναι ότι οι άνθρωποι που θα ζουν χωρί καθαρό νερό θα είναι 3,5 εκατομμύρια και δεν θα είναι μόνο σε φτωχέ χώρε και στη Σλοβακία όπου έχουμε αποθέματα υδάτων που όμως μολύνονται από βακτηρίδια ή από άλλες χημικές ουσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στις χώρες μέλη ότι δεν δρούν επαρκώς για να προστατεύσουν το νερό και μιλάει και για οικονομικά συμφέροντα επιχειρήσεων που εξαιτία τους δεν λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές για νερό ε, ποιότητας. Ξέρουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, ε, κάτι το οποίο συνεισφέρει σε ευρύτερε αλλαγές. Υπάρχει μετανάστευση, οπότε σίγουρα πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα. Συνάδελφε Μιράντα, για 1,5 λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το νερό είναι ένα δικαίωμα και είναι ένα κοινό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Κύριε Επίτροπε, ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει αυτό το δίκαιο και το δικαίωμα έτσι όπως το αναγνωρίζει ο ΙΕ και έτσι όπως έχουν κάνει χώρες όπως είναι η Βολιβία. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Στην Ευρώπη πρέπει να φροντίσουμε να προσφέρουμε ε, καθαρό ποιότητας πόσιμο είδωρ. Η Υπηρεσίε ίδρυυση πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να διασφαλιστεί η οικουμενική πρόσβαση στο νερό στην Ευρώπη. Αυτή η έκθεση όμως δεν συνάδει με τους αρχικούς στόχους που είχαμε. Δυστυχώς τα συμφέροντα παρεμβαίνουν και δεν καταφέρνουμε να έχουμε πραγματικά ε, πρόσβαση σε καθαρό νερό όπως θέλαμε, όπως γίνεται στην Ισπανία ή κι αλλού, που καταπατάτε αυτό το δικαίωμα στο νερό, στο καθαρό νερό για τους ανθρώπους και τα ζώα. Και ξέρω γιατί μιλάω, γιατί στη χώρα μου που έχει τόσα ποτάμια Κοστίζει πάρα πολύ το νερό, το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Οπότε περιορίζεται η πρόσβαση των πολιτών στο πόσιμο είδωρο, κάτι το οποίο είναι πολύ κρίμα. Συνάδελφε Φορέντσα, για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα καταψηφίσουμε την έκθεση Νταντέν. Είναι ένα κείμενο που πιστεύω ότι είναι πραγματικά δεν είναι παρκές και που προδίδει ε, το σκοπό του Κοινοβουλίου να βελτιώσει το κείμενο και να και και ένα από αυτό το Συμβούλιο. Είναι ένα κείμενο που δυστυχώ ε, παιδινώθηκε. Ο στόχο ήταν απλούστατο: να θυγαμιστούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με το αίτημα τη πρωτοβουλία των πολιτών, το right to water ή όπως είπε και ο ΙΕ, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό και αυτές οι υπηρεσίες του νερού να είναι καθολική δικαίωμα και να μην λαμβάνεται υπόψη το κέρδος και αγορά. Αλλά βλέπουμε μόνο μια σειρά ομών συστάσεων, απλών συστάσεων στα κράτη-μέλη. Σε άλλε εκθέσει δεν υιοθετήθηκαν επαρκεί παράμετροι, ούτω ώστε να συγκρατηθεί η ρήπανση των υδάτων από επικίνδυνε ουσίε που παράγουν οι βιομηχανίε, ε, όπω είναι οι ουσίε φας Φωσφορού ουσίε, εγώ θα καταψηφίσω. Το λέω σε εκατομμύρια Ιταλού πολίτε που ψήφισαν για ένα δημοψήφισμα για το δημόσιο νερό. Το οφείλω και στι γυναίκε, ε, στι μητέρε των παιδιών που ασθενούν και επίση και στου πολίτε που υπέγραψαν την πρωτοβουλία Right to Water. Η κυρία Ντορνάνο, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, οι ενδοκρινικοί διαταράχτες βρίσκονται παντού, στα ποτάμια, ε, στο νερό της βρύση λοιπόν, αυτό τελικά διαταράχουν το ορμονικό σύστημα αυτέ οι ουσίε και δημιουργούν φυσικές ανομαλίες συμπεριφορά και αναπαραγωγικέ. Λοιπόν, είχαν γίνει τρει κυβερνητικέ μελέτε που αφορούν το νερό, τι βρύσει στο νερό και τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Οι ενδοκρινικοί διαταράχτε είναι το ίμιση των παρασιτοκτόνων που είναι περισσότερο παρόντα. Η φύση των υδάτων ποικίλει ανάλογα με τι διάφορε χώρε και η εθνική κλίμακα είναι πιο κατάλληλη από ότι η ευρωπαϊκή αντιμετωπιστεί το θέμα. Όμως διαφωνώ με την τοποθέτηση του συγκητού όσον αφορά το αιτιολογικό. Αυτή η θέση προσπαθεί να ρεχιστοποιήσει τους κινδύνους αναφερόμενος σε έλλειψη επιστημονικής συνένεσης. Το ίδιο αφορά και την έρευνα για τα μικροπλαστικά που είναι απλώς είναι ένα πρώτο αρχικό στάδιο. Ζητώ συγγνώμη ότι η υγεία των ε, Γάλλων δεν είναι κάτι που είναι διαπραγματεύσιμο. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μάντελ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντω ισχύει ότι έχουμε δύο εκατομμύρια συμπολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό στα νοικοκυριά του. Είναι παιδιά εδώ, είναι ηλικιωμένοι. Συμμερίζομαι το στόχο ότι όλοι οι συμπολίτε μα στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν καθαρό νερό διότι αυτό θα σήμαινε ότι η Ευρώπη θα γινόταν η πρώτη ήπειρο όπου όλοι έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Θα ήμασταν πρωτοπόροι. Αλλά αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τι βελτιώσει τι οποίε επιφέραμε εμεί στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, η πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικέ ρυθμίσει και υπερβολική γραφειοκρατία. Γιατί το νερό στα περισσότερα μέρη είναι ήδη καθαρό. Δεν επιτυχάνουμε κανένα στόχο έτσι. Αντίθετα, αυξάνεται το κόστο για τα νοικοκυριά για όσους καταναλώνουν ε, νερό. Γι' αυτό και πάλι θα καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ο στόχος μπορεί να είναι σωστός, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε στην επόμενη θητεία από την αρχή σε αυτό το θέμα, για να επιτύχουμε καθαρό νερό για όσους δεν το έχουν ήδη. Υπάρχουν διάφορες παράλογες ε, παράμετροι που δεν προτείνονται καν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα πρέπει να φτιάξουμε ακόμη άλλες εγκαταστάσεις καθαρισμού πολλά ε, μέρη δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό θα καταψηφίσω αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να εργαστούμε όπω και στο παρελθόν περισσότερο για να επιτύχουμε πραγματικά του στόχου μα, Ούτω ώστε όσοι χρειάζονται και ακόμη δεν το έχουν, να έχουν στο μέλλον καθαρό νερό. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε Τσόφολη, για 1,5 λεπτό έχετε το λόγο. Δαμιάν, ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλούμεθα να επιβεβαιώσουμε την ψηφοφορία μα επ' αυτής τη σημαντικής για το δικαίωμα στο πόσιμο νερό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επικαιροποιήσει μετά από πάνω από 20 χρόνια για καλύτερα να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και για μια σωστή μετάβαση προς μια οικονομία κυκλική για να μειωθεί η σπατάλη του νερού και η παραγωγή πλαστικών αποβλήτων. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτε σχεδόν δύο εκατομμύρια από αυτού μα το ζήτησαν αυτό με την πρωτοβουλία του, για να εγγυόμεθα σε όλου, σε όλου το δικαίωμα στην πρόβαση την καθολική στο πόσιμο νερό. Ένα δικαίωμα ανθρώπινο πρωταρχικό που πρέπει να το εγγυηθούμε και όχι μόνο να το προωθήσουμε. Είναι θεμελιώδες ότι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφορίες ακριβείς και σαφείς όσον αφορά το είδωρ που βγαίνει από τη βρύση τους. Και όσον αφορά τη διαφάνεια, χαιρετίζω, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη μεγάλη ρήπανση από τα πφάς, από τις φωσχοριούχες ισίες που στην περιοχή του Βένετου στην Ιταλία έλαβε χώρα και περίπου αφορά περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες που έχουν ένα επίπεδο τέτοιων των ε, ε, δοκρινικών διαταρακτών εκατοντάδες φορές πάνω από τα όρια δεν είχαν, δεν είχαν προβλέψει οδηγίε όρια για αυτέ τι ουσίε. Όμω τώρα έχουν θεσπιστεί τα όρια, αλλά πρόκειται για όρια που είναι πολύ υψηλά. Θα πρέπει να φτάσουμε σε τιμέ κοντά στο μηδέν, όπω μα ζητούν οι πολίτε από το Βένετο και υπό το φω πρόσφατη γνωμοδότηση τη ΕΦΣΑ, που μείωσε το όριο των δόσεων των, ημερι... των καθημερινών που είναι ανοιχτέ στο αίμα. Ευχόμαστε το επόμενο κοινοβούλιο, στο επόμενο κοινοβούλιο και η Ιταλική κυβέρνηση εντό του Συμβουλίου και το Συμβούλιο και οι χώρες του Συμβουλίου που θα πρέπει να πάρουν οριστική απόφαση να καθορίσουν όρια που θα είναι κοντά στο μηδέν. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Τόμασιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα επίτευγμα η πρόσβαση στο νερό που δυστυχώς είναι κάτι που το παίρνουμε σαν δεδομένο. Κι όμως υπάρχουν νέες προκλήσεις, νέες προϋποθέσεις μπροστά μας. Είμαι από μια χώρα που έχει βέβαια πάρα πολλές πηγές ύδατος, αλλά γι' αυτό θέλω να σχολιάσω ότι πρέπει να τηρείται το πνεύμα της επικουρικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ελάχιστε προδιαγραφές ποιότητας. Ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Συνάδελφε Ροντρίκες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε είναι ανθρώπινο δικαίωμα το νερό και είναι και αναγκαίο για τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να βρίσκεται σε, στα χέρια ιδιωτών ούτε οι υποδομές γύρω από το νερό. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλικία, από όπου προέρχομαι εγώ, ε, έχουμε ποτάμια τα οποία έχουν ε, μολυνθεί από μεγάλα έργα που έγιναν για αυτοκινητοδρόμους, για παράδειγμα, υψηλής ταχύτητας και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε δεν είναι αποτελεσματικά για να σταματήσει αυτή η μόλυνση. Υπάρχουν ε, και άλλα σχέδια τα οποία γεμίζουν όλο και περισσότερο τα ποτάμια μας με ρηπογόνες ουσίες. Επίσης υπάρχουν και σταθμοί που υποτίθεται ότι είναι για ε, το καθαρισμό των υδάτων αλλά που στην ουσία ε, μολύνουν τα ποτάμια. Και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρνει καμία αντίρρηση. Δεν γίνεται έτσι να έχουμε καθαρό πόσιμο νερό. Ευχαριστώ συνάδελφε Γκαμπίου. Σχεδόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση που κάνουμε για την οδηγία για το πόσιμο νερό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί πρόκειται για την μοναδική πρωτοβουλία πολιτών που κατάφερε να προχωρήσει με πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές από τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ανησυχούν για αυτό το ζήτημα. Άρα η πρόσβαση στο νερό και η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται καλά και να τηρούμε επίσης και το στόχο 6 των ε, βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Είναι κάτι που ζητούν οι πολίτες μας. Και όταν μιλάμε για πρόσβαση, αυτό έχει να κάνει και με τα κοινωνικά δικαιώματα, που στο σημείο 20 ε, μιλούν για την πρόσβαση σε καθαρό νερό. Πρέπει λοιπόν, οφείλουμε να εγκρίνουμε την οδηγία αυτή, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε και έναν άλλο στόχο που έχει να κάνει με τα απόβλητα. Όταν έχουμε καλύτερη ποιότητα στο νερό που παίρνουμε από τη βρύση, θα καταφέρουμε να αποφύγουμε την κατανάλωση νερού σε πλαστικά μπουκάλια. Καλύτερη ποιότητα λοιπόν, καλύτερη πρόσβαση κυρίως για τους πιο ευάλωτους, για αυτούς που είναι στο περιθώριο και περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές όταν πρόκειται για το λογαριασμό που τους έρχεται στο σπίτι για το νερό και να βελτιωθούν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Πρόεδρε, συμφωνώ με τα λόγια του Πρόεδρου Γιούνκερ όταν ε, μιλούσε για την κατάσταση πραγμάτων στην Ένωση, που είπε ότι οι σημερινοί και οι μελλοντικοί πολίτες αξίζουν μια Ευρώπη που να προστατεύει τις προδιαγραφές της ζωής τους. Αξίζουμε μια Ευρώπη η οποία να μας ενισχύει, η οποία να βοηθάει και να προστατεύει. Τέλος, ευχαριστώ και συγχαίρω τον κύριο Νταντέν για το έργο του όσον αφορά αυτό το φάκελο. Όμως είναι κρίμα που παρά τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι χώρες μέλη δεν κατάφεραν να θεωρήσουν προτεραιότητα αυτό το ζήτημα και θα μείνουν οι διαπραγματεύσει για την επόμενη θητεία. Κρίμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ, συνάθε Ζωρίνιο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ και 20 χρόνια μιλάμε για το πόσιμο νερό και την ποιότητά του Μιλάμε για νερό ποιότητας που βέβαια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει. Τώρα η αναθεώρηση αυτή απορρέει από την πρώτη πρωτοβουλία πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών που προχώρησε όπου είχαμε 1,5 εκατομμύριο υπογραφές όσον αφορά την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε καθαρόν ναι, πόσιμο είδωρ. Θέλουμε λοιπόν μέτρα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε καθαρό νερό στους δημόσιους χώρους και το πόσιμο ίδρυ να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της επιστημονικής κοινότητας για το θέμα. Υπάρχουν πολλά θετικά που μπορούμε να υπογραμμίσουμε. Η μείωση της συγκέντρωσης ε, ουσιών όπως είναι ο ε, Όρια επίσης όσον αφορά τους εδοκρινικούς διαταράχτες βελτίωση των ε, διαδικασιών ε, για να αποφεύγουμε τα μικροπλαστικά, ελεύθερη πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα στο νερό της βρύσης. Επίσης, κυκλική οικονομία που συνεισφέρει στο να μειωθούν τα πλαστικά μπουκάλια. Όμως πάμε ακόμα πιο μακριά η πρόσβαση στο νερό και η μείωση των μικροπλαστικών δεν είναι τα μόνα θέματα. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στις φιλοδοξίες των πολιτών. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Φερέιρα. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αυτή η πρόταση που τροποποιεί την οδηγία για, την, ε, για το είδωρο για ανθρώπινη κατανάλωση έχει θεμελιώδη σημασία αυξάνει, αυξάνει συγγνώμη, όμως ε, το κόστος ε, της ε, χρήσης του νερού και θα το πληρώσουν οι καταναλωτές. Και επίσης αυξάνει το κόστος για τον έλεγχο της ποιότητας και δημιουργεί δυσχέρειες για τη δημόσια παροχή ύδατος, προωθεί την ιδιωτική παροχή ύδατος και ε, επιβάλλει περιορισμούς που δεν θα επιτρέψουν κυρίως για τις μικρές ε, εταιρείε παροχής ύδατος που λειτουργούν υπό την τοπική αυτοδιοίκηση στη λειτουργία τους. Πρέπει λοιπόν να αντικαταστήσουμε τον έλεγχο από τις δημόσιες αρχές από τον λεγόμενο αυτοέλεγχο. Στην ουσία είναι επικές με τις ιδιωτικές εταιρείε. Η πρόταση αυτή σημαίνει πιο ε, ακριβό νερό, λιγότερο ασφαλές και χειρότερης ποιότητας. σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει υποταγή στις μεγάλες ε, πολυεθνικές εταιρείες ε, που σχετίζονται με το νερό. Ευχαριστώ κυρία Σουίτσα για δύο λεπτά. Χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό οι πολίτες. Σύμφωνα με νέα ερεύνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, μόνο 40% των ευρωπαϊκών ποταμιών, λιμενών και των παρακτήων υδάτων πληρούν τις περιβαντικές προδιαγραφές ε, που βρίσκονται στην οδηγία περιδάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι σαφές τα περισσότερα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να συμμορφωθούν με τις επιταγές των οδηγιών ούτω ώστε στο μέλλον να έχουμε επαρκεί ποσότητε ποιοτικού νερού που θα παρέχονται για τι ανθρώπινε ανάγκε και το περιβάλλον. Η παρούσα οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ και ισχύει για 20 χρόνια χωρί σοβαρή αναθεώρηση Γι' αυτό το λόγο καλωσορίζω τις προσπάθειες ε, του εισηγητού και της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος να προσαρμοστούν οι προδιαγραφές για την ποιότητα του ποσίμου νερού ε, με βάση των πλέον προσφάτων επιστημονικών πορισμάτων για να υπάρχει ανταπόκριση σε νέα προβλήματα όπως είναι η αλλαγή του κλίματος. Για μία ακόμη φορά θέλω να τονίσω όλος ιδιαίτερος το πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρώτη πρωτοβουλία των πολιτών για το δικαίωμα στο είδωρ πάνω από 1,8 εκατομμύρια πολίτες υποστήξαν το δικαίωμα σε καθαρό ποιοτικό πόσιμο νερό. Είναι η ελάχιστη προδιαγραφή που πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ισχύει. Ο ΙΕ το έχει τονίσει και το έχει προωθήσει αυτό. Στην πατρίδα μου, την Κροατία, έχουμε αρκετό νερό, αλλά αυτή η πηγή, αυτός ο πόρος πρέπει να διαφυλαχθεί ως κοινό αγαθό. Χρειάζεται υπεύθυνη διαχείριση και χαίρομαι που σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα των πολιτών στο πόσιμο νερό. Επίση, υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προσπάθειε που καταβάλει για τη βελτίωση τη υγεία των πολιτών, αλλά λυπάμαι που ακούω ότι αναβάλλεται η απόφαση όσον αφορά αυτό το έγγραφο για την επόμενη θητεία. Ελπίζω, ε, καλωσορίζω όμω επίση ε, την εφαρμογή τη αρχή επικουρικότητα και στην επόμενη θητεία ελπίζω να καταφέρουμε βρούμε λύση. Συνάδελφε, πιετικά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάνουμε ένα βήμα, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό